παρακολούθηση τη κατάσταση εκ του και θα κινητοποιήσει την παροχή συνδρομής αν και εφόσον καταστεί αυτό απαραίτητο. Σα ευχαριστώ. Έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος για το τέλο τη συζήτηση. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε, η ψηφοφορία θα γίνει αμέσως μετά το πέρασα της συζήτηση και για τα δύο επόμενα θέματα. Το επόμενο είναι η Καμπότζη και ιδιαίτερα η περίπτωση του Σαμ Ρέινση. Ο πρώτος ομιλητής είναι η κυρία Σάκε. Δύο λεπτά κυρία Σάκε. Ευχαριστώ. Ο Σαμ Ρέινσι που είναι μέλος του Κοινοβουλίου στην Καμπότζη. Μόνο και μόνο γι' αυτό έγιναν απόπειρε δολοφονίες από το κυβερνό κόμμα ε, και του επιβλήθηκε μια δωδεκάμινη δωδεκαετής ποινή φυλάκισης. Δεν, δεν αρέσει στην κυβέρνηση το γεγονό ότι ο Σαμ Ρέινσι καταγγέλει τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τι περιπτώσει διαφορά. Μην ξεχνάμε ότι εμεί είμαστε ο μεγαλύτερο δωρητή βοήθεια στην Καμπότζη και θα πρέπει να βασίζεται αυτό στο σεβασμό από την Καμπότζη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 2006 ο Σαμ Ρέινσι έλαβε ένα βραβείο ε, για την υπεράσπιση τη ελευθερία. και υπερασπίζεται τις αρχές που υπερασπιζόμαστε κι εμείς. Ε, κάνουμε έκκληση στις αρχές της Καμπότζης να εφαρμόσει τις σύστασεις του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Καμπότζη. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ρωμέβα Ιρουέντα. Ευχαριστώ. Όπως... Νομίζω πως ε, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος στην ε, Καμπότζη, νομίζω πως δικαιούμεθα να ζητήσουμε από τις αρχές αυτής της χώρας να κάνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις και να δημιουργήσουν ένα δημοκρατικό κράτος με κράτος δικαίου που θα βασίζεται στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Αλλά πρέπει επίσης να καταπολεμήσουν την ενδυμική διαφθορά, τη μαζική αποδάσωση που οδηγεί σε εκτοπισμούς, την αρπαγή γης και τη βιομηχανία του σεξοτουρισμού να μειωθεί η ατιμορρησία και να οδηγηθούν ενώπιος δικαιοσύνης όσοι κάνουν όλες αυτές τις δραστηριότητες. Επίσης, η ελευθερία της πολιτικής έκφρασης είναι κάτι το αναγκαίο, αλλά πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να πούμε πως ανησυχούμε από την δίωξη και την καταδίκη σε δεκαετή κάθερξη του αρχηγού της αντιπολίτευσης Σαμ Ρέινσι με κατηγορίες που θεωρεί συμβολικές και πολιτικές. Είναι ανισχυτικό το ότι ακόμα αν επιβεβαιωθούν από δευτεροβάθμιο δικαστήριο αυτές οι κατηγορίες δεν θα μπορέσει να είναι υποψήφιος στις επόμενες ε, εκλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρωμέβα Ιρουέδα, η Βερονίκ Δεκαϊζέρ. Κύριε Πρόεδρε. Αυτό το κατεπήγον ε, ε, επικεντρώνεται στην αφιλεγόμενη πολλές φορές προσωπικότητα του σαν Ρέινση, αλλά θα πρέπει να ξεχνούμε ε, το πραγματικό δημοκρατικό διακύβευμα, γιατί ο Σαμ Ρέινση είναι φιλελεύθερος, είναι αντιπολίτευση κατά του Προέδρου Σαμ και ήδη καταδικάστηκε σε 18 μήνες και το 2006 έλαβε αμνηστία επειδή υποτίθεται ότι ήταν ηθικός αυτούργος μιας δολοφονικής απόπειρας με χειροβομβίδα. Σήμερα καταδικάζεται για μια συμβολική πράξη, μετέθεσε ουσιαστικά τα, τα φυλάκια της, των αφιλεγόμενων συνόρων μεταξύ Βιετνάμ και Καμπότζης και υποτίθεται παραποίησε τοπογραφικούς χάρτες. Είναι σαφές ότι αυτό που θέλουν οι αντίπαλοι του είναι να τον εμποδίσουν να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές του 2013, ενώ είναι ο αρχηγός του δεύτερου κόμματος ε, αντιπολίτευσης σε αυτή τη χώρα. Έχουμε ένα πολύ τεταμένο πολιτικό κλίμα, επίκειται εκλογές, γίνονται κάποιοι πολιτικοί χειρισμοί και ελιγμοί, αλλά υπάρχει και μια αυταρχική συμπεριφορά της κυβέρνησης. Εκτός από το Sam έχουμε και εκπροσώπου μη κυβερνητικών οργανώσεων που διώκονται. Έχουμε την ε, βουλευτή Ναμού Σόσουα, που καταδικάστηκε σε δυσφήμιση σε βάρος του Πρωθυπουργού. Έχουμε την, το δημοσιογράφο Χανκ Σάκρα που κρατήθηκε επί εννέα μήνε επειδή κατήγγειλε τη διαφορά στο περιβάλλον του Αντιπρόεδρου Σοκάν και ούτω καθεξής. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι ε, είμαστε σημαντικό χορηγό βοήθεια στην Καμπότζη και έχουμε και συμφωνίε συνεργασία που προβλέπουν ότι θα πρέπει να τηρούν τη θεμελιώδη ελευθερίε. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω εφαρμογή εκτάκτου σχεδίου ανθρωπιστική βοήθεια για του πληθυσμού που έχουν πληγεί εξαιτία τη κρίση στο κατασκευαστικό και κλωστοφονταριοκό κλάδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Δεκάιζερ. Ο Τσάρλ Στάνοκ. Ε, η Καμπότζη στα χαρτιά είναι πλουραλιστική δημοκρατία όμως, ανθρωπιστικές οργανώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις λένε ότι ε, οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν εκφοβισμούς ε, και βία. Η δικαιοσύνη είναι αδύναμη και υφίσταται πολιτικές πιέσεις. Η κυβέρνηση όμως κλείνει τα μάτια ε, στην παράνομη αρπαγή γης, στην παράνομη λιωτόμηση και στην λαιλάτιση των φυσικών πόρων. Ο ο αρχηγός της αντιπολίτευση, ο οποίος είναι αυτοεξόριστος στη Γαλλία, ε, καταδικάστηκε ρήμην σε 12 ετή ποινή φυλάκισης ε, για το θέμα της συνοριακής ε, διαφοράς με το Βιετνάμ. αυτό το ψήφισμα είναι επίκαιρο και θα πρέπει να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση ε, τους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσει επίσης τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλιώς θα, θα στυλιτευθεί ε, στη διεθνή κοινότητα ως παρείας η Καμπότζη. Ευχαριστώ. Κυρία Μακοβέ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ένας ηγέτης αντιπολίτευσης καταδικάστηκε ερήμην σε δεκαετή κάθερξη Βεβαίως η δίκη του δεν ήταν αμερόληπτη και είχε πολιτικά κίνητρα. Παρόμοιες καταδίκες μελών της αντιπολίτευσης είναι διαδεδομένες και δείχνουν πως δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην Καμπότζη και έτσι εμποδίζονται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα όπως το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και τη δίκαιη δίκη. Αντιτίθεμε στην καταδίκη του Σαμ και άλλων οι οποίοι προσπαθούν να εκφράσουν ελεύθερα την ε, γνώμη τους και ζητά από την κυβέρνηση της χώρας να σταματήσει αυτή την τυραννία. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την Καμπότζη να οδηγηθεί στη δημοκρατία και να μην εφαρμόζει επιλεκτικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ζητά από την Κομισιόν να υπενθυμίσει την Καμπότζη να μην χρησιμοποιήσει νέου κανονισμούς για τη ΜΚΟ για να περιορίσει την κοινωνία των πολιτών και την αντιπολίτευση. Ευχαριστώ. τώρα οι ομιλητέ ξενομοτή ομάδων, η κυρία Εσαϊά για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Στην Καμπότζη υπάρχει μια αυταρχική κυβέρνηση και με αυτοαρχικό τρόπο διευθύνει τη χώρα. Οποιοςδήποτε εκφράζει κριτική, οποιοδήποτε δικαστής, οποιοδήποτε δημόσιος υπάλληλος φημώνεται. Το ξέρουμε γιατί πολλοί καταδικάστηκαν μόνο και μόνο γιατί υπερασπίστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος ε, δωρητής βοήθειας στην Καμπότζη, ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας ε, και θα πρέπει να γίνει κάτι με τις πολυάριθμες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στην Καμπότζη το πρώτο άρθρο, το άρθρο 1 τη συμφωνία συνεργασίας με την Καμπότζη που τονίζει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. θα πρέπει η βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να είναι προπόθεση τη χορήγηση βοήθεια στην Καμπότζη. Κυρία Κρέτσου. Ευχαριστώ. Είναι αλήθεια ότι μια καταδίκη σε 12 φυλάκιση αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μία απόδειξη του αυταρχισμού που δεσπόζει στην πολιτική ζωή της Καμπότζης. Επίσης, ε, αποκλεισμό του από την Εθνική Βουλή, επειδή η βουλευτική ασυλία ανακλήθηκε τουλάχιστον τέσσερις φορές και τέσσερις ε, οπαδοί του κόμματος έχασαν τη ζωή τους σε μία επίθεση με χειροβοβίδα, μας ε, βάζουν υποψίες για το πόσο αρνητική είναι η κατάσταση στην Καμπότζη και πώς οι πολιτικοί του αντίπαλοι προσπαθούν να τον εμποδίσουν να συμμετέχει στις εκλογές του 2013. Όλα αυτά υπονομεύουν τη δημοκρατία στην υποτιθέμενη δημοκρατία της Καμπότζης. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να σταματήσει τις πολιτικές διώξεις και να ζητήσουμε από την ύπατη εκπρόσωπο για τις εξωτερικές υποθέσεις να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό μέσο για να ζητήσει από την κυβέρνηση να σεβαστεί πραγματικά τη δημοκρατία στη χώρα. Κυρία Ευχαριστώ, κύριε. Χέφνερ για του πράσινου 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Καμπότζη είναι μια εξαιρετικά όμορφη χώρα με μεγάλη ιστορία, αλλά η ιστορία αυτή έχει και φρικτές πτυχές, ιδιαίτερα επίκαιρες. Εξαφανίζονται άνθρωποι, συλλαμβάνονται χωρίς λόγο. Υπάρχει πολύ υψηλή διαφθορά, παράνομη υλοτομία, αρπαγές γης και αυτοί οι οποίοι ασκούν κριτική σε αυτή την κατάσταση τους τσιμπάνε από το δρόμο και στείνουν εικονικές δίκες στις βάρους τους. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πούμε πως πρέπει να υποστηρίξουμε τον Σαμ Ρέιντσι ήδη από το 1995 απομακρύνθηκε από το Κοινοβούλιο, κατάφερε να επανεκλεγεί, έχει επιζήσει πάρα πολλών επιθέσεων ε, σε προεκλογικές ε, εκστρατείες. Σε μία από αυτές σκοτώθηκαν 80 άτομα. Εγώ είχα την ευκαιρία να τον επισκεφτώ και είναι ένας συναρβαστικός άνθρωπος, ε, μαχητής της ελευθερίας και τώρα με, ισχνά, με ένα ισχνό κατηγορητήριο έχει συλληφθεί. Όποιος βεβαίως φυλακίζει τον επικεφαλής αντιπολίτευσης, ε, φυλακίζει και ένα υψηλό ποσοστό κατοίκων της χώρας ε, του που τον ψήφισαν. Όποιο εμποδίζει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης να κατέβει στις εκλογές, εμποδίζει την δημοκρατία και τα δικαιώματα των πολιτών. Δεν πρέπει να το δεχτούμε αυτό και απευθύνω έκκληση στην Κομισιόν να τηρήσει ιδιαίτερα το άρθρο 1 της Συμφωνίας Συνεργασίας με την Καμπότζη που αναφέρει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως προϋπόθεση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπιέλαν τώρα, εκ μέρους της ομάδας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ. Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ δύο φορέ στην Καμπότζη πριν από δύο χρόνια για πρώτη φορά σε μια αποστολή παρατήρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των ε, βουλευτικών εκλογών και τη δεύτερη φορά πριν από έξι μήνε. Η Καμπότζη είναι μια χώρα που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με ραγδαίου ρυθμού ενώ από οικονομική άποψη. Το ίδιο όπως και άλλες χώρες εκείνη της περιοχή του κόσμου. Δυστυχώ παρά την ραγδαία οικονομική ανάπτυξη, δεν έχουμε αντίστοιχο γρήγορο εκδημοκρατισμό. Δεν έχουμε μια γνήσια δημοκρατία στην Καμπότζη. Γιατί ε, δεν έχουμε ούτε ισχυρή αντιπολίτευση, ούτε ισχυρά μέσα μαζική ενημέρωση ούτε ισχυρέ με κυβερνητικέ οργανώσεις. Η ε, καταδίκη του κυρίου Σαμράνση, που είναι η δεύτερη καταδίκη του ηγέτη της αντιπολίτευσης, και είναι μια προσπάθεια να εμποδιστεί να συμμετέχει σε επόμενες βουλευτικές εκλογές, γιατί είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στη χώρα του. Αυτή η απόφαση λοιπόν ει βάρο του είναι πολύ σημαντική, γιατί πολλές φορές ε, μέλη του, των ΧΜΕΡ έχουν ε, κριθεί και καταδικαστεί στην Καμπότζη. Δυστυχώ ε, η στάση αυτή τη κυβέρνηση δεν συμβάλλει στην αποστα... στη σταθεροποίηση τη περιοχή και θα πρέπει η κατάσταση να διαθετηθεί με πολιτικά μέσα και όχι με δικαστικέ αποφάσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μπασέσκου, στα πλαίσια τη διαδικασία ε, Catch the Eye. Θέλετε να μιλήσετε λοιπόν, κυρία Μπασέσκου. Αν θέλετε, τώρα είναι η ώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι αξιοθρήνητο που το Δικαστήριο της Καμπότζης χρησιμοποιεί τη σύλληψη ως μέσο εκφοβισμού των μελών της αντιπολίτευσης και των αντιφρονούντων. Αυτοί που είναι τα πρώτα θύματα είναι οι ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλοι όσοι είναι υπέρ της ελευθερίας έκφρασης. Θεωρώ ότι οι κατηγορίες ε, εναντίον του Σαμ Ρέινσι έχουν ένα πολιτικό χαρακτήρα, πιο πολύ παρά δικαστικό. Καταδικάστηκε σε μια ποινή φυλάκισης 12 ετών μετά από μια συμβολική χειρονομία που έκανε. Διαμαρτυρήθηκε για τον τρόπο που σχεδιάστηκαν τα σύνορα με το Βιετνάμ. Νομίζω ότι η πραγματική αιτία όμω τη φυλάκισής του είναι η θέληση τη κυβέρνηση να μην του δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία για τι επερχόμενε εκλογέ του 2013. Ε, θα έπρεπε να κάνουμε μια έκκληση στην κυβέρνηση τη Καμπότζη, να σεβαστεί τι δεσμεύσει τη για τη δημοκρατία. Ο Σαμ Ρέινς είναι ο βασικός εκπρόσωπος αντιπολίτευσης και θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επανέλθει στο Κοινοβούλιο της Καμπότης το συντομότερο δυνατόν και να σταματήσει αυτό το σύστημα, το σύστημα το μόνο κομματικό το οποίο είναι επιζήμιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ο επόμενος ομιλητής. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Η απόφαση εις βάρος του Σαμ Ράινσι, η καταδίκη του δηλαδή σε δεκαετή κάθριξη για την υποθέμενη αυτή απάτη ε, αποτελεί αιτία για σοβαρή ανησυχία για την εξαρτησία της δικαιοσύνης ε, σε αυτή τη χώρα. Η κυβέρνηση πραγματικά σκοπεύει να εμποδίσει την αντιπολίτευση να κάνει οτιδήποτε. Και βεβαίως του στερεί την ελευθερία τους. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις ε, στην Καμπότζη από όταν επικρατούσε τρομοκρατία και έχουν αληφθεί κάποια βήματα για να γίνει ένα δημοκρατικό κράτος. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαφυλάξουμε αυτές τις εξελίξεις στην Καμπότζη και σε άλλες χώρες περιοχής. Ευχαριστώ. Τώρα βλέπω τον κύριο Πρέντα. Έχετε λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η περίπτωση του Σαμερένση, όπως αναφέρθηκε και είναι χαρακτηριστική γιατί αυτός ο άνθρωπος καταδικάστηκε δύο φορές, την πρώτη φορά ε, για δύο χρόνια φυλάκισης και τη δεύτερη φορά για άλλα δέκα. Κατηγορήθηκε για παραποίηση εγγράφων και παραπληροφόρηση. Όπως όμως είπαν πολλοί, ήταν μια πολιτική διαμαρτυρία ε, και στόχος της απόφασης ήταν να εμποδιστεί από τους αντιπάλους και να συμμετέχει σε επόμενες εκλογές. Ο Σάμ ουσιαστικά καταδικάστηκε για πολιτικούς λόγους. Καταδικάστηκε ερήμην μετά από δύο ακροματικές διαδικασίες που έγιναν και κλεισμένο των θυρών και δεν σεβάστηκαν τις αρχές της ε, δικονομίας και της ε, διεξαγωγής της δίκης δίκης. Δεν ήταν ο μόνος ε, αρχηγός αντιπολίτευσης ή ο μόνος αντιφρονών που υπέστη πολιτική δίωξη. Όπω είπαν πολλοί, μπορούμε να στηριχθούμε στι συμφωνίε συνεργασία που έχουμε συνάψει με την Καμπότζη και να ζητήσουμε από τη χώρα αυτή να σεβαστεί τι υποχρεώσει τη ε, για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κύριο Πάσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε. Η Καμπότζη, όπως και άλλες, χώρε, χώρες, ε, εκεί διεξάγεται ένας αγώνας για την πολιτική εξουσία και ο αγώνας αυτός παίρνει διαστάσεις ζωής και θανάτου. Οι αρχές στην Καμπότζη έχουν τη διάθεση να εξαφανίσουν τους αντιπάλους τους, να τους φυλακίσουν. Οι αρχές προσπαθούν να ξεφορτωθούν το Σάμ Rainsy γιατί είναι κίνδυνος για αυτές. Γιατί ίσως ε, ενσαρκώνει την ελπίδα για μια πολιτική αλλαγή. Ίσως θα μπορούσαμε να παρέμβουμε και να ζητήσουμε από την κυβέρνηση της Καμπότζης να σταματήσει τη δίωξη των πολιτικών αντιπάλων της θα πρέπει να δοθεί ευκαιρία στο, στο Sam να συμμετάσχει στον εκλογικό αγώνα. Νομίζουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήταν πιο επιτυχής από τις προηγούμενες προσπάθειές τους. Θα πρέπει να ασκήσουμε πολιτική πίεση στην Καμπότζη, να τη ζητήσουμε να αλλάξει συμπεριφορά και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για ελεύθερες εκλογές και πολιτικές διαδικασίες στη χώρα. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Έχω Εφτά σχέδια ψηφίσματος για το τέλος της συζήτησης αυτής. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, θέλω να δώσω το λόγο στην, Επίτροπε, στην Επίτροπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές που συμμετείχαν στην συζήτηση για την Καμπότζη. Πράγματι εκεί πέρα η κατάσταση είναι ανησυχητική. Είχαμε ειλικρινείς συνομιλίες με τους ε, συνομιλητές μας από την Καμπότζη τελευταία φορά στις Βρυξέλλες 8 ε, Οκτωβρίου και ιδιαίτερα για τη μεταχείριση της αντιπολίτευσης. Το γεγονό πως ο Σαμ Ρέιντζι αναγκάστηκε να ζητήσει καταφύγιο στη Γαλλία είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης η οποία επιδεινώνεται. Το ίδιο ισχύει και για την ανάμειξη δικαιοσύνης πολιτική και την δίωξη ανθρώπων που θα έπρεπε να έχουν ε, βουλευτική ασυλία. Οπότε η Εθνική Εθνοσυνέλευση θα μπορεί πλέον να λειτουργεί ως ε, μέρος για την ελεύθερη έκφραση απόψεων, ούτε και τα μίμια. Από την άλλη, η Καμπότζη αποδέχτηκε στην περιοδική επιθεώρηση του ΟΗΕ όλες τις παρατηρήσεις. Επίσης, βλέπουμε πως υπάρχει ένας νέος ποινικό κώδικας και νόμους κατά πολέμης διαφθοράς, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν και βέβαια πρέπει να υπενθυμίσουμε στην Καμπότζη τις παρατηρήσεις των εκλογικών παρατηρητών στο παρελθόν. Επίσης ε, πρέπει να καταστεί αποτελεσματική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνει η κυβέρνηση και να συστήσει και ένα κοινό φόρουμ με οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Η Καμπότζη παραμένει μια φτωχή χώρα Πολλά μπορούν να γίνουν για να συνεχιστεί η πρόσφατη οικονομική ανάπτυξη χωρίς να αυξάνονται οι ανισότητες στην κοινωνία. Αυτό πρέπει να συμπεριλάβει μεταρρύθμιση των κανόνων ιδιοκτησίας γης και να σταματήσουν οι μία η φόρες πρακτικές ε, δασοκομείας συμπεριλαμβανομένης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων. Το να τιμωρήσουμε την κυβέρνηση ή να μειώσουμε το επίπεδο των επαφών δεν θα ωφελήσει σε τίποτα τους φτωχότερους και θα ενθαρρύνει εκείνους οι οποίοι μόνο στα λόγια υποστηρίζουν τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει υποκατάστατο του υπομονετικού διαλόγου. Εάν δεν θεωρηθούμε σοβαρό εταίρο στην ανάπτυξη τη χώρα, δεν θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε τα γεγονότα. Υπάρχουν όμω πολλά τα οποία μπορούμε να κάνουμε στην Καμπάτη σε, ό, σε, Καμπότη, σε όλα τα επίπεδα. Από το γραφείο του Πρωθυπουργού μέχρι την κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τι πρωτοβουλίε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη ισότητα ενώ θα συνεχίσουμε να ζητάμε μια πραγματική πλουραλιστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, πιο ελεύθερο τύπο και ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επίτροπο. Τελειώνει η συζήτηση για την Καμπότζη, για την περίπτωση του Σαμ Ρέινσι. Θα ψηφίσουμε ως Νούπο, Αλλά πριν να περάσουμε στην ψηφοφορία, έχουμε ακόμα ένα σημείο να συζητήσουμε για το Βόρειο Κάφκασο και κυρίως την περίπτωση του Όλεγ Ορλόφ. Η συζήτηση θα ξεκινήσει με την παρέμβαση της κυρίας Χαουτάλα. Πρόεδρε, αυτό το ψήφισμα για την κατάσταση στο Βόρειο